La seduta è Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Comunico. Να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αριθμός ψηφισάντων 737. Λευκά, άκυρα 73. 662 ψηφίσαντες. Απόλυτη πλειοψηφία για την εκλογή είναι οι 332 ψήφοι λοιπόν. Οι υποψήφοι έλαβαν τις εξής ψήφους. Η κυρία Κέλλερ, 133 ψήφους. Η κυρία Ρέγκο, 42 ψήφους. Ο κύριος Ασόλη, 325 ψήφους και ο κύριος Ζαχραντήλ 162 ψήφους. Επειδή κανένα υποψήφιο ε, δεν έλαβε απόλυτη πλειοψηφία ψήφων, περνάμε σε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οι νέες υποψηφιότητες εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρες οι υποψηφιότητες της πρώτης ψηφοφορίας. Υπάρχει κάποια παρατήρηση? Έλαβα λοιπόν τις ακόλουθες υποψηφιότητες. Κυρία Σκάκελερ. Κυρία Σύρα Ρέγο. Ο κύριος Ντάβιτ Μαρία Σασόλη. Και ο κύριος Γιάννη Βάχαρης. Αν δεν υπάρχουν νέες υποψηφιότητες, θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στις 40. Ε, διακόπτεται η συνεδρίαση, θα συνεχίσουμε στις 12 παρα 20, 11.40. Il Presidente. La seduta è ripresa. Επαναλαμβάνεται η Σύνοδος. Πριν προχωρήσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία, ήθελα να ξέρω αν όλοι οι ψηφολέκτες ε, είναι παρόντες και έχουν λάβει θέση. Κύριε Γιάρ, παρακαλώ να καθίσετε στη θέση σας. Κύριε Γιάρ. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρόεδρε Μπούζεκ. Πρόεδρε Μπούζεκ. Κύριε Τάλερ, είστε εδώ. Είστε εδώ, κυρία Τάλερ. Κυρία Τάλερ. President Buzek is here. Πρόεδρε Μπούζακ, είστε εδώ. President Buzek is, is coming. Έρχεται ο πρόεδρος Μπούζακ. Μόλις φτάσει ο πρόεδρος Μπούζακ, είναι θα ξεκινήσει η διαδικασία. Happy birthday, President Buzek. Χρόνια σας πολλά, κύριε Μπούζεκ. Χρόνια πολλά. Προχωρούμε στη δεύτερο, στο δεύτερο γύρο ψηφοφορία. Καλώ του ψηφολέκτε να λάβουν τι θέσει του κοντά στι κάλπε και θα, θα αναλάβουν μετά το τέλο τη ψηφοφορία. Έχετε λάβει του φακέλου με τα ψηφοδέλτια, άρχεται η ψηφοφορία.